donc tu es d'accord pour Colleghi, buongiorno. Eh, cominciamo. Καλημέρα σα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε αμέσω. Καθίστε, σα παρακαλώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε αυτή την ε, πρωινή συνεδρίαση για τη διαφθορά. Ο τίτλο είναι «Η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση στο θέμα τη διαφθορά. Θα ακούσουμε το Γενικό Διευθυντή της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Στεφανό Μανσερβίση, που θα μας μιλήσει για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό κατά της Διαφθοράς με συγκεκριμένη αφορά στην έκθεση κατά της Διαφθοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν μετά την παρουσίαση του κυρίου Μανσερβίση θα ακούσουμε το Γενικό Γραμματέα του Γκρέκο, του Βόρφαν Γκράου, που θα μας μιλήσει για την ανάγκη αύξηση της διαφάνεια και την καταπολέμηση τη διαφορά από τη σκοπιά του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, θα έχουμε 15 λεπτά για την παρουσίαση του κάθε προσκεκλημένου και κατόπιν θα ανοίξουμε τη συζήτηση δίνοντα το λόγο καταρχήν στου συντονιστέ, κατόπιν στους κύριου βουλευτέ ε, και κατόπιν ε, στους προσκεκλημένου για να απαντήσουν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε Αλφάνο και σας ευχαριστώ, ε, ευχαριστώ την Επιτροπή σας ε, για την πρόσκληση, για αυτή τη συνεισφορά σε αυτή την ε, πολύ ευαίσθητη εποχή για την Ευρώπη. Θα μιλήσω σε αγγλικά, νομίζω ότι είναι καλύτερα για όλους. Και πάλι σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστώ για το έργο σας που είναι μια πρόκληση που πρέπει να συνεχίσουμε γιατί νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε κυρία θέματα που σχετίζονται στενά με την προσπάθεια της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν δεν είναι μεμονωμένη. Βρίσκεται ε, στο εσωτερικό της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την ε, οικονομική κρίση, τη χρηματοπιστωτική κρίση, την χρήση της απασχόλησης και την κρίση της αξιοπιστίας των θεσμών. Νομίζω λοιπόν ότι το πρώτο θέμα είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και η πρωτοβουλία που πρέπει να αναλάβουμε είναι να το θέσουμε σε ένα πλαίσιο να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην οικονομία και στην αγορά και στους θεσμούς. Υπάρχουν κάποιοι υποστοκομμένοι παράγοντες. Ε, σύμφωνα ε, με έγγραφα γνωρίζουμε τη σχέση μεταξύ της διαφθοράς ε, και των μεγάλων δημοσιονομικών ελλημάτων. Ήδη κάποια χρόνια ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι η διαφθορά κλέβει από την ελληνική οικονομία 20-30 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω δωροδοκιών και αυτό αντιστοιχεί στο 12% του ΕΠ. Σύμφωνα με το Global Financial Integrity. 160 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν στην Ελλάδα λόγω παράνομης φυγής κεφαλαίων μέσα σε μια δεκαετία μέχρι το 2009. Επίσης, μια σημαντική έκθεση του Ιταλικού Ελεκτικού Συνεδρίου εντόπισε περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε έτος, περίπου το 4% του Ιταλικού ΑΕΠ, ότι είναι το κόστος της διαφθοράς. Αυτό ε, που επιβεβαιώθηκε το 2012 και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην Ιταλική οικονομία. Για να πούμε λοιπόν κάποια ε, αριθμητικά στοιχεία τα οποία είναι γνωστά Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτό σχετίζεται με τις προσπάθειες της οικονομικής μεταρρύθμισης στην Ευρώπη. Στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020, επίσης, εξετάζουμε το συσχετισμό μεταξύ της αντίληψης της διαφθοράς και της οικονομικής ανάκαμψης και το συμπέρασμα ήταν ε, ότι η διαφθορά ε, επηρεάζει ε, την επίτευξη των στόχων τους Ευρώπης 2020. Και αυτό σαφώς υπολογίζεται όχι μόνο στην ποσότητα των χρημάτων που χάνονται, αλλά αποστοικοποιείται και με πολιτικούς όρους. Γιατί τελικά τι έχει νόημα εδώ η σημασία των δικτών που πολύ συχνά παραγωνίζονται. Συνεχώς εμείς ε, εξετάζουμε το ΑΕΠ, την αύξηση της παραγωγικότητας, όλα αυτά φυσικά είναι σημαντικά, αλλά υπάρχουν και άλλοι δείκτες ε, που αφορούν ε, την οικονομική ανάκαμψη και την θεσμική μεταρρύθμιση και είναι σημαντικό πώς είναι το κράτος δικαίου, καλή διακυβέρνηση και ο έλεγχος της διαφθοράς. Αυτοί είναι δείκτε που είναι λιγότερο προφανής ή παρουσιάζονται λιγότερο από το αλλά νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικοί. Γνωρίζετε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχει κι άλλο ένα νούμερο, 120 δισεκατομμύρια ευρώ που χάνονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, στα 27 κράτη-μέλη λόγω της διαφθοράς στις δημόσιες προμήθειες, σύμφωνα με μελέτες περίπου 20-25% ε, της αξίας ε, των συμβάσεων χάνεται λόγω της διαφθοράς και φαντάζομαι ότι ε, είναι πολύ χαμηλότερα αυτά τα νούμερα από ό,τι στην πραγματικότητα γιατί ξέρετε είναι εύκολο να ε, σε κάτι που φαίνεται κάπως ξεκάθαρο όμως έχουμε θέμα έλλειψης εμπιστοσύνης στην πραγματική οικονομία ποιε δραστηριότητε χάνονται, γιατί υπάρχει αστάθεια και υπάρχει και διαφθορά. Επίση, υπάρχουν και κάποιε ενδιαφέρουσε πτυχέ ε, που παρουσιάζει το Ευρωβαρόμετρο σε σχέση με τη στάση και την αντίληψη των Ευρωπαίων προ τη διαφθορά. Δημοσιεύτηκε φέτο το Φεβρουάριο. Τρει από τους τέσσερις πολίτε συνεχίζουν να θεωρούν μεγάλο πρόβλημα τη διαφθορά στη χώρα τους και περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι το επίπεδο τη διαφθορά στη χώρα του αυξήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Και ένα πιο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο για τη διαφθορά μας έδειξε ότι 40% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι μια πολύ στενή σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικής συνεισφέρει στη διαφθορά. Αυτό είναι πολύ αυστηρή κρίση γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον οικονομικό αντίκτυπο, αλλά και με τον πολιτικό αντίκτυπο. Αν η ίδια φθορά δεν έχει μόνο οικονομικό αντίκτυπο, ε, που ήδη είναι καταστροφικός, ε, αλλά ουσιαστικά υποσκάπτει την αξιοπιστία της δημοκρατίας, ε, αυτό δημιουργεί πραγματικά απειλή στην κοινωνία μας, όχι μόνο από οικονομική σκοπιά, αλλά και στην αξιοπιστία των πολιτικών μας και των δημοκρατικών θεσμών. Και ανοίγει ε, ουσιαστικά το χώρο για να επικρατήσουν άλλες πολιτικές δυνάμεις. Έχοντας λοιπόν αυτό κατά νου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται τώρα για την παραγωγή ενός μηχανισμού, τη δημιουργία ενός μηχανισμού κατά της διαφθοράς για να βοηθήσουμε την προσπάθεια των κρατών μελών κατά της διαφθοράς. Ε, θα εργαστούμε λοιπόν επί αυτής της έκθεσης εντοπίζουμε κάποιους τομείς που θα καλύπτει η έκθεση αυτή και θα ήθελα να πω Ξέρετε, θα είμαστε ταπεινοί, δεν θέλουμε να επανεφεύρουμε τον τροχό, ούτε πιστεύουμε ότι θα αποκαλύψουμε εντελώ νέους δείκτες ή γεγονότα. Θέλουμε να προσθέσουμε, διότι να καταρχήν ότι αναλαμβάνει η Ευρώπη τη δική της ευθύνη σε αυτό, έτσι λοιπόν να ε, παγιώνουμε ορισμένα στοιχεία, και εντοπίζουμε ποιες δράσεις θα αναλάβουμε. Και δεύτερον, αυτό σχετίζεται με την αξιοπιστία του οικοδομήματο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, ο βαθμός ε, της ολοκλήρωσης είναι σαφής. Αυτό σχετίζεται με την αξιοπιστία αυτών των οργανισμών και η διαφθορά είναι στο κέντρο αυτού και επίσης ε, λαμβάνουμε δράσεις για να μειώσουμε τους κινδύνους ε, που θα μπορούσαν να προκύπτουν από προβλήματα και να μας οδηγήσουν σε κρίση. Έτσι λοιπόν η έκθεση κατά της διαφοράς, καταρχήν ε, αποτελεί μια έκθεση, μια, ένα εγχείρημα εξυγίανσης θα ασχοληθούμε με κάποια οριζόντια θέματα και σε κάποια ζητήματα που αφορούν πιο συγκεκριμένα κάθε κράτος μέλος. Ε, όπως σας είπα, ενοποιούμε κάποιες πληροφορίες που έρχονται από διάφορες πηγές. Ε, έχουμε και κάποιους μηχανισμούς παρακολούθησης όπως ο Γκρέκο, το Ούνκα, Κοσά και θα χρησιμοποιήσουμε ε, ε, και δεδομένα που έχουμε και από άλλες πηγές όπως η Transparency International και άλλες αξιόπιστες οργανώσεις που εργάζονται επί αυτού του φαινομένου, του παθολογικού φαινομένου της οικονομίας και της πολιτικής που είναι διαφθορά. Η Κομισιόν στο πλαίσιο αυτό θα κάνει και κάποιες συγκεκριμένες ε, συστάσεις προκειμένου να προτείνει κάποιες οδούς στα κράτη-μέλη έτσι ώστε τουλάχιστον ε, να καταδειχθούν οι δυναμίες τους. Θέλουμε να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες το επίπεδο της διαφθοράς των χωρών τους, αλλά ακόμη το πιο σημαντικό είναι γιατί εμείς ε, δεν θέλουμε να δεκτυλοδείξουμε κάποιον, απλώς ε, θέλουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να συμμετέχουν περισσότερο οι πολίτες. Η ιδέα μα είναι να αναφέρουμε συγκεκριμένε δράσει που θα μπορούσαν να αναλυφθούν προκειμένου να ανοίξουμε τι οδού για συζήτηση, για, για κριτική αλλά και για δράση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και επίση η πρόθεσή μα είναι να αναφέρουμε και κάποιε επιτυχημένε περιπτώσει, γιατί δεν είναι όλα σάπια. Έχουν αναλυφθεί κάποιε πρωτοβουλίε που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ω σημείο αναφορά από άλλου. Τώρα, πότε Ήδη είχαμε μια αρχή στην περσινή ανακοίνωση που την είχαμε συμπεριλάβει εκεί. Τώρα εργαζόμαστε με αυτό. Σχεδιάζουμε να εκδώσουμε αυτή την έκθεση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του 2013. Συζητήσαμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διαφθορά που από 17 μέλη και εργάζεται από τον Ιανουάριο για το, επί του θέματος αυτού. Έχουμε ένα δίκτυο ε, τοπικών ε, ερευνητών που αναλύουν τα δεδομένα Όλοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι, συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, άτομα από την κοινωνία των πολιτών και ερευνητέ. Ε, δεν έχουμε δηλαδή εδώ την διακυβερνητική προσέγγιση, γιατί θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε χαμηλότερο επίπεδο στη συζήτηση. Επίσης, ε, έχουμε ε, κάποια σημεία που θα επικεντρωθούμε και το μεγαλύτερο θα είναι οι δημόσιες ε, συμβάσεις. Όπως σας είπα, χάνεται μέχρι και το 25% της αξίας των συμβάσεων και εργαζόμαστε προκειμένου να εστιάσουμε στις δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να εντοπίσουμε ποια είναι τα κύρια ζητήματα, τα κύρια αδυναμίες στο σύστημα. Ήδη προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά μέσω της αναθεωρημένης οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις το Δεκέμβριο του 2011 Επίσης, να λάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες, όπως αυτή που είναι υποσυζήτηση, σε ό,τι αφορά την οδηγία ε, για τα, και την κατάσχεση των εσόδων που προέρχονται από εγκληματικέ δραστηριότητες. Ξέρετε, πολλές φορές ε, δεν είμαστε ε, δεν κατορθώνουμε να γνωστοποιήσουμε το τι κάνουμε, όμως ε, η καταπολέμηση της διαφοράς, η καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος, η καταπολέμηση δεδομένων που ε, καταστρέφουν την οικονομία μας και καταστρέφουν την, την δημοκρατία, αυτή είναι η βασική έννοια, ότι επιτιθέμεθα κατά όλων αυτών και βλέπουμε όλες τις μεταλλάξεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και αυτό είναι το τμήμα του εγχειρήματο. Δεν θέλουμε λοιπόν να διαχωριστούμε εμεί από τα κράτη-μέλη σε μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά και σε όλο ένα, ε, και μια, μια πιο συνεκτική αρχιτεκτονική πολιτική διακυβέρνηση και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, θα εξετάσουμε και τι ακριβώ συμβαίνει στο δικό μα επίπεδο. Και Προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποια είναι τα βασικά θέματα. Τώρα, καλή διακυβέρνηση και πολιτικέ ε, κατά τη διαφθορά, όπω σα είπα, αυτά αποτελούν τμήμα των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη σύσταση ε, που υλοποίησε η Κομισιόν σε κάποια κράτη-μέλη στο τέλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, είχαμε εκεί συγκεκριμένες συστάσεις προς συγκεκριμένα κράτη-μέλη, προκειμένου να τονιστούν ακριβώς προβλήματα που έχουν σε αυτό το τομέα. Και φυσικά αυτό συνοδεύει και άλλες προσπάθειες ε, που κάνουμε σε άλλους τομείς. Δεν είναι εύκολο και επαναλαμβάνω. Δεν ε, θέλω τώρα να ε, καυχηθώ εδώ ότι κάνουμε κάτι επαναστατικό. Απλώς προσπαθούμε να βρούμε ποιοι είναι οι κύριοι δείκτες και τα αριθμητικά στοιχεία για να δούμε πόσο σημαντικά είναι αυτά για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αξιοπιστία της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών. Και θέλουμε αυτή την έκθεση η οποία ε, εξετάζει τι συμβαίνει. Θέλουμε να παρουσιάσουμε τι τάσει αλλά και συγκεκριμένε πληροφορίε, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί καλύτερα. Πρόκειται για μια διαδικασία λοιπόν, την οποία θέτουμε σε κίνηση και θα είναι ζωτική συνεργασία μας ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω και της δημιουργίας αυτής της ειδική επιτροπής. Ε, όπως ε, εργάζεστε εδώ, θέτετε το σκηνικό. Δηλαδή, ουσιαστικά απευθύνεστε σε όλους τους θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορούν να ληφθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από νομοθετική σκοπιά, από πολιτική σκοπιά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Και νομίζω ότι το κοινό μας έργο τις επόμενες εβδομάδες είναι πολύ σημαντικό. Να είστε επικριτικοί, να είστε συμμαχοί μας, εμείς πάντως το είμαστε συμμαχοί σας, προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό το σημαντικό έργο που έχουμε ενωπιών μας. Και σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, διότι Ιδίως τονίσατε την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα ε, και Ιδίω σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή ε, Νοσή ε, και την οικονομική κρίση. Το παρακαλώ τώρα τον κύριο Ράου να ε, παρουσιάσει το θέμα του που είναι η ανάγκη στην Ευρώπη να αυξήσουμε τη διαφάνεια. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Είναι μεγάλη ε, χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι σε αυτή την σημαντική ε, συνάντηση σχετικά με την καταπολέμηση της ε, ε, διαφθοράς. Καταρχήν όμως ε, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για τον οργανισμό μου, την Κρέκο, που καταρτίστηκε το 1999 για να παρακολουθεί την εφαρμογή των έξι των έξι διατάξεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και ε, σε αυτές περιλαμβάνεται ε, και ε, η σύμβαση για το ποινικό δίκαιο σχετικά με την διαφθορά. Τώρα έχουμε στην ομάδα αυτή 49 κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Καταρτίζονται αξιολογήσεις σχετικά με την ανάλυση της της νομοθεσίας και το αποτέλεσμα είναι ότι η Γκρέκο μπορεί να αναφερθεί και να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις ανά χώρα βάσει μίας εκθέσεως αξιολόγησης. Αλλά αυτό είναι απλούστατα ένα σκέλος της εργασίας μας. Το άλλο σκέλος είναι η αξιολόγηση επιπτώσεων η οποία μετά από κάποιο χρόνο ε, αξιολογεί εάν τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν από τη χώρα για να εφαρμοσούν οι συστάσεις επαρκούν και σε τέσσερους γύρους αξιολογήσεως η Γκρέκο έχει εξετάσει διάφορα θέματα δηλαδή ε, με τα, ε, ε, πολλά θέματα αλλά μεταξύ αυτών θα αναφερθώ εις ε, την ανεξαρτησία και την εξειδίκευση και τα διαθέσιμα μέλη, μέτρα για τα, τους εθνικούς οργανισμούς να προλάβουν και να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, την εφαρμογή της νομοθεσίας ε, της ε, της ε, διαφθοράς και την ορισμένα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την σταθερότητα των ε, δημοκρατικών θεσμών. Σε ένα μήνα θα έχουμε την πρώτη έκθεση για την ε, Σλοβενία, ε, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο και θα ήθελα να σας πω σχετικά με την διαφάνεια ότι είναι ο σαφής αντίποδας στην ε, διαφθορά και σε πολλά θέματα η ευαισθητοποίηση, η κατάργηση φραγμών στην πληροφόρηση, η εφαρμογή υποχρεώσεων αποκαλύψεως και ενίσχυση ελεγχών ε, μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχω επιλέξει περιοχές που είναι σημαντικές για τον οργανισμό μας στην Κρέκο. Καταρχήν ε, χρειάζεται διαφάνεια στην δημόσια διοίκηση και στις ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λήθος για την πρόληψη της διαφθοράς. Σημαίνει ότι η οργάνωση, η λειτουργία και η διαδικασία λήψεως αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την καταπολέμηση της διαφθοράς και να εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ε, διαφάνεια. Ε, η Γκρέκο κάνει μία έκκληση κατά τρόπον ώστε να διευκολυνθεί και ε, να υλοποιηθεί η εύκολη πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση των, σχετικά με τους δημόσιους οργανισμούς. Όσον αφορά την ομοθεσία πληροφόρησης πρέπει να είναι απλή και όχι περίπλοκη περιλαμβάνοντας προϋποθέσεις που θα εμποδίσουν την πρόσβαση σε πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, εάν πρέπει πάντοτε οι πολίτες να ζητούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ή να εξηγήσουν για ποιο λόγο τις θέλουν δεν θα διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία. Για μας λοιπόν η ελεύθερη πρόσβαση στις, στην πληροφόρηση ε, πρέπει να είναι ο κανόνας. Το δεύτερο μου παράδειγμα είναι ότι έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς οι οποίοι αναφέρουν υπόνοιες ε, ε, διαφθοράς αυτούς δηλαδή που μαρτυρούν τους ε, ατάκτους whistleblowers ε, ε, για να αποφευθεί η συγκάλυψη. Το whistleblowing λοιπόν είναι ε, αυτή η αναφορά, είναι ένας τρόπος για να αυξηθεί η η διαφάνεια ε, και να υπάρξει μεγαλύτερη ακαιρεότητα και να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να καταπολεμήσουμε και το οργανωμένο έγκλημα. Οπότε οι καλοί πίστεως ε, ε, που μαρτυρούν μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να, και πρέπει να προστατεύονται από αντίπεινα. Έτσι υπάρχει ένας μηχανισμός εφαρμοστικός με τον, μέσω του οποίου ερευνούνται τα παράπονα της, των αντιπίνων και ε, μπορεί να υπάρξει επανόρθωση. Βέβαια υπάρχουν διάφορες ε, κατηγορίες ε, ερετών ε, ή δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι προστατεύονται από τις προσφυγές και γι' αυτό χρειάστηκε να υπάρξουν σαφείς κανόνες σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της διαφθοράς χωρίς να υπάρχουν αντιφάσεις <clears throat> που, διότι η διαφάνεια είναι η βάση της δημοκρατίας. Η Γκρέκο λοιπόν έχει ε, ε, συστήσει σε μία σειρά κρατών η οι ε, κατάλογοι ή οι κατηγορίες αυτών οι οποίοι προστατεύονται από ασυλία να μειωθεί και αυτό ιδίως όσον αφορά τους βουλευτές και τις ε, διαδικασίες της ε, άρσεως της ασυλίας. Όσον αφορά την ε, ε, εξέλιξη και τη σταδιοδρομία των δημοσίων ε, στελεχών που είναι πολλές φορές και καλυμμένοι και όπου υπάρχουν διάφοροι αρνητικοί παράγοντες χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και να εξασφαλίσουμε ότι η πρόοδος θα οφείλεται στην αξία τους ε, και θα γίνεται σωστή αξιολόγηση των υποψηφίων για προαγωγή. Ε, πέμπτον, ε, η διαφάνεια αυτή είναι βασική αρχή σχετικά με τα αντικρουόμενα. Δηλαδή, εάν δημόσια στελέχη πρέπει να ε, υποβάλουν ε, δηλώσεις σχετικά με τα περιουσιακά τους στοιχεία πράγμα το οποίο εφαρμόζεται όλο και ε, περισσότερο οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων όπως ο ανεξήγητος πλούτος θα μπορέσουν να αποκαλυφθούν πιο εύκολα και κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρχει υπάρξει ένα επιπλέον βασικό όπλο κατά της διαφθοράς. Όσον αφορά τους ε, βουλευτές, ε, πολλές φορές ε, υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα τα οποία πρέπει να εξηγήσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και γι' αυτό χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια και δυνατότητα αποκάλυψης των στοιχείων ε, ιδίως όσον αφορά τις επαφές των βουλευτών με τρίτους που μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη των αποφάσεών τους. Ε, δεν πρέπει ε, να πρέπει να υπάρξουν συστήματα ηθικής και να προστατεύονται οι βουλευτές από τα παράνομα συμφέροντα. Τώρα όμως θέλω να αναφερθώ και στα πολιτικά κόμματα και στους, ε, στις προεκλογικές εκστρατείες ε, και έχει ε, πολλές φορές αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει επαρκής νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατιών. Χρειάζονται ε, πολλές φορές ε, να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν άμεσες δωρεές, δάνεια ε, και ε, χορηγίες οι οποίες ε, έχουν χρησιμοποιηθεί ε, για να παρακαμφθούν οι κανόνες που διέπουν τέτοιες χορηγίες και δωρεές. Σε ορισμένες χώρες δεν αναφέρονται και δεν αποκαλύπτονται οι δωρεές παρά μόνο εάν πρόκειται για πολύ μεγάλα ποσά. Και η νομοθεσία πολλών κρατών αγνοεί ε, την, ε, ε, την την τοπική αυτοδιοίκηση που μπορεί επίσης να είναι ευάλωτη σε τέτοιες περιπτώσεις αυτή η, αξιολόγηση της χρηματοδοτήσεως των πολιτικών κομμάτων ε, σημαίνει ότι ε, οι χώρες δεν έχουν κάνει όλες ισότιμες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν αυτές τις ατέλειες και σε ορισμένες χώρες υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά και δεν υπάρχει καμία εφαρμογή των συστάσεων για τη χρηματοδότηση των κομμάτων ε, και η συνολική τους ε, ε, ε, αντιμετώπιση έχει θεωρηθεί από την Γκρέκο σαν ε, γενικός ε, μη ικανοποιητική, πράγμα το οποίο μας δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Καταλήγοντας λοιπόν, η αύξηση της ε, ε, διαφανείας δεν ε, είναι η μαγική λύση για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, ούτε μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά στην πρόληψη. Ε, πρέπει να εξετάσουμε όλες τις ε, εναλλακτικές λύσεις και όταν πρόκειται ε, για ε, υψηλού βαθμού διαφθορά χρειάζεται στις χώρες αυτές να υπάρξει αντίστοιχη νομοθεσία. Ξέρουμε από το Ευρωβαρόμετρο ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της διαφθοράς στην Ευρώπη από ό,τι φανταζόμασταν. Άρα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία για να μπορέσει να νομιμοποιηθεί το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του και θα πρέπει η καταπολέμηση της διαφθοράς να τοποθετηθεί σε αυτό το γενικό πλαίσιο όχι μόνο για να βελτιωθεί το επιχειρησιακό περιβάλλον αλλά για να αμώσουν και οι δημοκρατικοί θεσμοί διότι όταν βλέπετε ότι οι ελάχιστοι προσέρχονται να ψηφίσουν στις εκλογές αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί πρέπει να αποκατασταθεί ε, το κύρος των πολιτικών και στα πλαίσια της εργασίας σας ενδεχομένως σας ενδιαφέρει να ακούσετε ότι ε, το ε, Συμβούλιο της Ευρώπης προσφέρει πρόκειται να καταρτήσει μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων για το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και ε, υπάρχει και η ιδέα το η λευκή βίβλος αυτή που θα καταρτιστεί να προτείνει ορισμένες ενέργειες του Συμβουλίου της Ευρώπης προς αυτή την κατεύθυνση και ε, ελπίζω ότι θα υπάρξει συνεργασία με την τωρινή σας και μελλοντική σας εργασία. Ε, ένα τελευταίο θέμα. Νομίζω ότι μία από τις πιο βασικές ε, προκλήσεις ε, είναι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για μας. Ιδίως ε, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην εργασία της Επιτροπής Γκρέκο και θεωρούμε ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι δεδηλωμένη αλλά πρέπει να ενισχύσουμε την, το αποτελεσματικότητα των αμοιβαίων προσπαθειών μας και χρειάζεται να συσφιχθεί η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να αποφευχθούν επικαλύψεις και ασάφειες οι οποίες δεν θα ήταν προς όφελος αυτής της πολιτικής στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι θα βρεθεί μια ικανοποιητική ε, λύση και ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, η Γκρέκο θα μπορέσουν να συνεργαστούν επικοδομητικά για να συμβάλλουν στην εφαρμογή των συστάσεων της Γκρέκο πέραν της ασκήσεως της αξιολογήσεως την οποία προβαίνεται τώρα για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τη διαφθορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Ε, στην ε, παρουσίασή σας επισημάνατε επανειλημμένα αυτό που κατά την άποψή μου είναι ε, το κομβικό σημείο, δηλαδή η χρηματοδότηση των κομμάτων, των προεκλογικών εκστρατιών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πολλές φορές δεν διέπονται από διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν σίγουρα αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη από πλευρά των πολιτών απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει, υπάρχει μηδενική αν όχι η εμπιστοσύνη. Θα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων ε, και ξεκινάμε με ε, Ματιού, εκ μέρους του ΕΛΚ με την κυρία Ματιού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά, κύριε Γενική Διευθυντά, είμαι πολύ ικανοποιημένη που η Κομισιόν ξεκινά μια μελέτη για την διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι ότι θα περιοριστείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πάντως ε, είμαι πολύ ικανοποιημένη από το γεγονός αυτό. Αναφέρεται τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, ε, από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για ένα ε, νούμερο που δεν είναι πάγιο σταθερό και μιλήσατε και για την αξιοπιστία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ηθική, γιατί πρόκειται για κλοπή. Νομίζω ότι όταν μιλάμε περί κλοπής, ε, κατανοούμε πολύ περισσότερο περί ως πρόκειται. Όσοι είναι διφθαρμένοι είναι πολύ απλά κλέφτες. Και πρέπει η Κομισιόν να κάνει αυτή τη μελέτη. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και αναμένουμε την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να μας πείτε, αλλά ίσως είναι κάπως νωρίς και να μην έχετε δεδομένα αν αυτή η διαφθορά ή μειώνεται. Γιατί έχουμε κάποια κράτη-μέλη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως Κομισιόν κάνατε ήδη κάποιες προτάσεις ό,τι αφορά τη διαφθορά. Να μας πείτε λοιπόν αν σημειώνεται αύξηση ή μείωση στη διαφθορά και κυρίως από την κρίση του 2008. Αν η κρίση αυτή είχε αντίκτυπο στη διαφθορά και αν η διαφθορά σχετίζεται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό. Τώρα, κύριε Ράου, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, πολύ σημαντική και πλήρης. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όμως θα ήθελα να μην είχατε αναφερθεί στην χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές ε, και αυτό θα σήμαινε ότι ε, δεν είναι αρκετά αξιόπιστη πολιτική. Μην ξεχνάτε ε, ότι ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο ένα και χαμηλότερη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι διεφθαρμένα. Σε κάποιες χώρες, ε, όχι απαραίτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ απογοητευμένοι οι πολίτες από τους πολιτικούς τους που είναι διεφθαρμένοι όταν όμως εμείς ε, βλέπουμε ως ευρωβουλευτές ότι δυσκολευόμαστε να πείσουμε τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν. Δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι διφθερμένοι. Δεν λέω ότι όλοι ε, είναι ενάρετοι, αλλά πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί σε αυτά που λέγονται. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ο κύριος Νιούτον Ντάν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, δύο μιλητές γιατί αυτά που μας είπαν ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχήν απευθύνομαι προς την Επιτροπή. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντίγραφο ε, της ομιλής σας, γιατί αναφέρετε πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Εγώ προσπάθησα να τα καταγράψω όλα, αλλά θα ήταν χρήσιμο να μου τα δώσετε κι εσείς σε γραπτή μορφή. Δεύτερη ερώτηση. Έχω την εντύπωση ε, ότι η διαφάνεια είναι το κλειδί. Το είπαν αυτό και οι δύο μιλητές. Η διαφάνεια βαρόμετρο της παγκόσμιας διαφθοράς, το παγκόσμιο βαρόμετρο διαφθοράς, μοιάζει αυτό με το ευρωβαρόμετρο και πολλά από τα πορίσματα είναι παρόμοια. Εδώ βασικά ζητάμε από τους ανθρώπους να μας πούν τη γνώμη τους και να μας πούν ε, πόσο μεγάλο θεωρούν το πρόβλημα της διαφθοράς στη χώρα τους. Στο τελευταίο βαρόμετρο συνειδητοποιήσαμε εξή. Βασικά πήραμε συνεντεύξει ε, από ανθρώπους σε 86 χώρε ε, σε 24, σε 24 ευρωπαϊκές χώρες και τους ρωτήσαμε αν εμπιστεύονται τους θεσμούς του, ε, αν πιστεύουν ότι μπορούν να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Εδώ έχουμε τις 24 ευρωπαϊκές χώρες που συμπεριλάβουμε σε αυτή τη μελέτη και να σας δώσω ένα παράδειγμα για μία από, την ε, ερω... μία από τις ερωτήσεις. Μία από τις ερωτήσεις ήταν πώς άλλαξε το επίπεδο διαφθορά στη χώρα σας, τι πιστεύετε. Και από όλε ε, τις περιφέρειες ε, στον κόσμο, η Ευρώπη ήταν αυτή όπου είχαμε το 73% των πολιτών να απαντούν ότι θεωρούν ότι το πρόβλημα της διαφθοράς έχει αυξηθεί. Μια άλλη ερώτηση που θέσαμε στους πολίτες ήταν σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι οι θεσμοί πλήττονται από τη διαφθορά. Και εδώ οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι τα πολιτικά κόμματα και τα κοινοβουλία τίνουν περισσότερο προς τη διαφθορά σε σύγκριση με άλλους θεσμούς. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το βαρόμετρο που αφορούσε την άποψη των πολιτών, όμως διερευνήσαμε τι συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα για να συμπληρώσουμε την έρευνά μας και να πετύχουμε το στόχο του να εξετάσουμε το πρόβλημα από διαφορετικές σκοπιές. Το 2011 δημοσίευσαμε μία έκθεση που λέγεται «Διαφάνεια στην εταιρική υποβολή εκθέσεων» γιατί Όσα ξέρουμε εμεί ω ΜΚΟ είναι ότι δημοσιεύουν εταιρείε. Μπορούμε λοιπόν να αξιολογήσουμε μόνο και να παρακολουθήσουμε τον κίνδυνο τη διαφθορά από τη σκοπιά των πληροφοριών που έχουν δημοσιεύσει οι εταιρείε. Και εδώ μεθοδολογία είναι ενδιαφέρουσα γιατί είδαμε την αποκάλυψη των πληροφοριών σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις. Καταρχήν, μια εταιρεία ανέφερε τα προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς, δηλαδή προγράμματα συμμόρφωσης σε ιστορικό επίπεδο, ιστορικούς κανόνες, για το πώς να αντιμετωπίζουν θέματα όπως η δωροδοκία, σύγκρουση συμφερόντων, δεύτερον, αποκάλυψη σε οργανωτικό επίπεδο. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο πληροφορίες σχετικά με την ε, διακυβέρνηση μιας πολυεθνικής, αλλά και πληροφορίες ε, σχετικά με τις θηγατρικές, ε, τα holding, τα κατοφυλάκια κτλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για μια πολυεθνική εταιρεία. Και η τρίτη διάσταση είναι η αποκάλυψη χρηματοοικονομικών πληροφοριών αναχώρα ή ανα Και αυτό σημαίνει τι πληρωμές ε, καταβάλει μια πολυεθνική όταν λειτουργεί στο εξωτερικό, δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, πόσες πληρωμές δικαιωμάτων καταβάλλονται σε κυβερνήσεις κτλ. Η μελέτη αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε πέρσι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα γιατί μας έδειξε ότι πολλές εταιρείες ε, δεν ε, προβαίνουν σε υποβολή εκθέσεων. Ε, ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιες ε, βελτιώσεις σε τομείς ε, όπως δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή, όπως στο πετρελαϊκό τομέα, στο τομέα των ορυχείων, το με το αερίου, όμως ιδίω ο τραπεζικός τομέας και ο χρωματοποστατικός τομέας δεν υποβάλλουν αρκετές εκθέσεις σε καμία από τις τρεις, στα τρία επίπεδα που μόλις σας ανέφερα. Εδώ βλέπετε ένα κατάλογο. Έχουμε βάλει στον κατάλογο αυτό τις εταιρείε. Και σημειώσαμε ότι για μια εταιρεία όπως η Στατόιλο ή η Rio όπου υπάρχει αρκετή πίεση προς αυτές από την κοινωνία των πολιτών για αποκάλυψη πληροφοριών και στις τρεις κατηγορίες, έχουν κάνει καλή δουλειά ενώ ως εταιρείε ε, βλέπετε στο κάτω μέρος ε, του καταλόγου έχουμε εταιρείε όπως ε, China Constructions, την Τράπεζα της Κίνας και άλλες τράπεζες στο κάτω μέρος του καταλόγου που δεν αποκαλύπτουν επαρκείς πληροφορίες και έτσι ώστε η κοινωνία και άλλοι υποπτικοί οργανισμοί να παρακολουθήσουν τι κάνουν. Τώρα για να αναφέρω και τα τρία επίπεδα Τη υποβολή εκθέσεων όταν ε, οι εκθέσει αναφέρουν να έχουν προγράμματα κατά της διαφθοράς. Εδώ η πλειονότητα των εταιριών κατά μέσο όρο υποβάλλουν κάποιες εκθέσεις. Όταν ε, υποβάλλουν εκθέσεις ε, σε σχέση με την ε, οργανωτική διαφάνεια. Έχουμε 45 από τις 105 εταιρείε ε, που υποβάλλουν καλές εκθέσεις. Όμως έχουμε πάρα πολλές εταιρείε που με τα βίας υποβάλλουν εκθέσεις και σε αυτή την τρίτη κατηγορία που μας ανησυχεί περισσότερο η διάσταση της υποβολής ένα χώρα. μας ανησύχησε ότι 41 από τις 105 εταιρείε έχουν Πολύ κακή επίδοση. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα της μελέτης ήταν ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας ε, έχει τις χειρότερες επιδόσεις. Τώρα, για να απομακρυνθώ από τον ιδιωτικό τομέα, θα πάω στο επόμενο τομέα. Κάναμε μία έρευνα μέσω των εθνικών μας γραφείων επιτόπου και εδώ θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Εργαστήκαμε πολύ ε, σκληρά. Έχουμε κάποιες ΜΚΟ στις χώρες διεύρυνσης που εργάζονται πολύ σκληρά, αλλά και σε πολλές όμορες χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Εδώ αξιολογείται η πρόοδος ε, των κυβερνήσεων από έτος έτος και έχουμε τη δημοσίευση αιτήσεων εκθέσεων κατά της διαφοράς ε, που χορηγούμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε εκεί να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στις αξιολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και ένα ακόμη σχέδιο, ένα ακόμη project που θέλω να τονίσω που υλοποίησε η Transparency International το είναι μελέτη του Συστήματος Εθνικής Ακαιρεότητας, NIS, σε 23 χώρες στην Ευρώπη. Το NIS βασικά είναι αυτό που αποκαλούμε μια ολιστική προσέγγιση έρευνας, όπου προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τις αδυναμίες ε, των ε, Συστημάτων ανακαιρότητα στις διάφορες χώρες. Εξετάζουμε τους διάφορους πυλώνες, ξεκινώντας ε, από το δικαστικό, το δημόσιο τομέα, την εκτελεστική εξουσία, τα πολιτικά κόμματα και προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν αδυναμίες. Γιατί υπάρχουν αδυναμίες, υποθέτουμε ότι μια χώρα έχει κακά στάνταρ διακυβέρνηση ε, και υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος διαφθοράς. Στην έκθεση αυτή που μόλις ολοκληρώσαμε, προσδιορίσαμε ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις ε, στην Ευρώπη Υπάρχουν κάποια σημαντικά ελλείμματα, κάποιες σημαντικές ελλείψεις, αλλά και κάποιες επασχόμενες πρακτικές που θα ήθελα να τονίσω. Επίσης, ε, το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ιστορικών Υποθέσεων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευχαριστούμε. Και εδώ έχουμε τις κύριες τάσεις που εντοπίσαμε στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθοράς, ε, τα περισσότερα νομοθετικά πλαίσια είναι καλά αναπτυγμένα. Το δεύτερο θετικό που είδαμε είναι ότι οι δημόσιες ε, δαπάνες, η επισκόπηση των δημόσιων δαπανών ε, γίνεται με ικανοποιητικό τρόπο στις χώρες με εξαίρεση της Ελλάδας, Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Ισπανία Βρήκαμε αδυναμίες ε, σε αυτούς τους θεσμούς και το τρίτο είναι η διαδικασία η εκλογική, η οποία είναι ευρούστη και με ξέρει στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ε, είδαμε να υπάρχει καλή επίδοση. Σε αυτές τις χώρες πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι σε όλη την Ευρώπη βρήκαμε έξι κυρίες αδυναμίες που ουσιαστικά συμπίπτει με όσα είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Είδαμε ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών ε, κομμάτων δεν έχει ρυθμιστεί επαρκώ σε όλη την Ευρώπη. Συστήνουμε λοιπόν να υπάρξουν καλύτεροι κανόνες σε όλη την Ευρώπη. Αλλά και σε ό,τι αφορά και τα ευρωπαϊκά κόμματα. Στην ομιλία του κ. Μπαρόσο για την κατάσταση της Ένωσης, ε, Αναφέρθηκε ότι υπάρχει μία μεταρρυθμίση που μόλις ξεκίνησε για τα ευρωπαϊκά κόμματα και εμείς νομίζουμε ότι αποκάλυψη πληροφοριών σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων είναι κάτι σκόπιμο. Γιατί ακόμη δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για τις δωρεές κυρίως. Το δεύτερο πρόβλημα που εντοπίσαμε ήταν ε, το lobbying και άσκηση πιέσεων Στι πρωτεύουσε της Ευρώπης αλλά και στι Βρυξέλλες. Πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά για να είναι πιο διαφανές ε, αυτό το lobbying και άσκηση πιέσεων. Ήδη εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε υποχρεωτικά μητρώα για τα λόμπι. Τώρα με τις νέες εξουσίες που απέκτησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ενθαρρύνουμε την ΕΚΤ να μπει και στο Μητρό Διαφάνεια σε ευρωπαϊκό γιατί πιστεύουμε ότι περισσότερες εξουσίες πρέπει να συνάδουν με περισσότερη λογοδοσία. Και θα πρέπει, και μάλλον προβλέπουμε να υπάρχει περισσότερη άσκηση πίεση στη Φρακφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενδυναμώσουμε το Μητρό Διαφάνεια που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτο, που εντοπίσαμε είναι ότι τα κοινοβούλια δεν ανταποκρίνονται στα ηθικά πρότυπα. Το είδαμε αυτό το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, αλλά και εδώ στι Βρυξέλλε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα νέο κώδικα δεντολογία. Αυτό ο κώδικα δεντολογία ε, είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, αλλά θα πρέπει και να εφαρμοστεί. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια κενά σε αυτό το κώδικα δοντολογία. Ε, το συζήτησα για κλεισμένο των θυρών. Ελπίζουμε ότι αυτή η συζήτηση να γίνει πιο δημόσια σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς ε, για τα δώρα και τη φιλοξενία και άλλες πτυχές. Ελπίζουμε ότι τη Συμβουλευτική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δοντολογίας επίσης θα ενδυναμωθεί. Τέταρτη αδυναμία, πρόσβαση στις πληροφορίες. Πέμπτο, υψηλό κινδύνος διαφθοράς και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Και έκτον, ε, καταγγελίες, whistleblowing. Αυτά είναι οι τομείς που εντοπίσαμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μιτερμάιερ. Τώρα ο κύριος Χρυσικός έχει το λόγο από το UNODC. Το φιλοξένησαμε και χθε, ήταν ο μιλητή μα και χθε και σήμερα θα μα μιλήσει για την αξιολόγηση τη κατάσταση τη διαφθορά και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σχετικά με την μέτρηση, τον εντοπισμό και τη μέτρηση της διαφθοράς και θα εμπνευστώ από σχόλια των προλαλισάντων. Η διαφθορά είναι ένα πολυσχεδές φαινόμενο και δεν μπορούμε να ε, εντοπίσουμε το φαινόμενο αυτό εάν δεν ε, ε, αποδεχθούμε ότι υπάρχει διαφορετική τυπολογία της διαφοράς και διάφοροι τρόποι και διάφορα περιβάλλοντα που πρέπει να εξεταστούν και να αναλυθούν αναλόγως του εθνικού περιβάλλοντος για να καταλήξουμε σε, έγκυρες, σε έγκυρα συμπεράσματα σχετικά με τη διαφθορά. Υπάρχει και πολυμορφία ε, θεσμικών οργανισμών που πρέπει να εξεταστούν για να λύσουμε το θέμα της διαφθοράς οπότε πρέπει να σας πω ποια είναι η προοπτική του οργανισμού UNODC δηλαδή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα από δύο σκοπιές καταρχήν από πλευράς του γενικού πλαισίου και δεύτερον ε, από πλευράς επιστημονικής ε, της ε, μετρήσεως της διαφθοράς. Το σημείο λοιπόν εκκινήσεώς μας σχετικά με το θεσμικό θέμα ε, των προτύπων είναι ε, η σύμβαση ε, του, των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της διαφθοράς που ψηφίστηκε το 2005 και ε, ο μηχανισμός αναθεώρησής της που καταρτίστηκε το 2009 για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι πολιτικές εναντίον της διαφθοράς ή στις εθνικές νομοθεσίες. Αυτό που είναι βασικό για αυτή τη σύμβαση είναι η αρχιτεκτονική του συστήματος και τα μέτρα που μπορούν και να προλάβουν την ε, διεθνή εγκληματικότητα και συνεργασία στα θέματα της διαφθοράς. Βλέπουμε τις διάφορες τυπολογίες της διαφθοράς όπου περιλαμβάνονται ε, διάφορα θέματα όπως παραδείγματος χάρη χρηματοδότηση ε, των πολιτικών κομμάτων, δημόσιες προμήθειες ενώ από πλευράς ε, εγκληματικότητος υπάρχει ένας εκτενής κατάλογος των ποινικών αδικημάτων που πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ελέγχονται και αντιμετωπίζονται εις ε, την ε, εθνική νομοθεσία για να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση. Ένα θέμα θεσμικό είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί είναι η αναθεώρηση των επιπτώσεων της ε, διαφθοράς μέσω καταλήλων μέτρων τα οποία θα αντιμετωπίσουν τα διάφορα αδικήματα που συνδυάζονται με τη διαφθορά και αυτά γίνονται από τον οργανισμό που εφαρμόζει την ε, σύμβαση ε, με μία τριπλή κίνηση καταρχήν να προωθήσει και να διευκολύνει και να αναθεωρήσει την εφαρμογή να προβεί σε συστάσεις και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμβαλωμένων το πιο βασικό, η δομή μάλλον της διάσκεψης αυτής των κρατών που συμμετέχουν στη σύμβαση εμφανίζεται στη διαφάνεια αυτή και βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες εργασίες ε, σχετικά με ε, την ε, πρόληψη της διαφθοράς με την τεχνική βοήθεια και ε, του ε, ε, εξέβρεση των πόρων που έχουν διασπαθιστεί και βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες παράμετροι και διάφορες διαστάσεις και στα πλαίσια αυτά και τα Ηνωμένα Έθνη και η Παγκόσμια Τράπεζα συνεργάζονται στην πρωτοβουλία για την ανάκαμψη των πόρων για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη και να βοηθήσουν τις εθνικές διοικήσεις να αναπτύξουν ένα καλύτερο μηχανισμό που θα εντοπίζει θα αναγνωρίζει και θα επαναπατρίζει τα προϊόντα των εγκληματικών ε, ενεργειών που έχουν ε, ε, ε, επενδυθεί ε, ή τοποθετηθεί στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν ο βασικός οργανισμός που επιβλέπει τις συνεχείς ε, ε, εκθέσεις και τις ε, αναθεωρήσεις της διαδικασίας κατά τρόπον ώστε ο μηχανισμός αυτός ο οποίος υιοθετήθηκε στην Τόχα το 2009 και βασίζεται ε, σε μία διαδικασία αναθεώρησης μεταξύ ομοτήμων υπάρχουν αναθεωρητές οι οποίοι εντοπίζονται και καθορίζονται ε, μέσω κλήρου και είμαστε τώρα στο, στον πρώτο κύκλο δηλαδή την εφαρμογή ε, των κεφαλαίων που αναφέρονται εις την ποινικοποίηση και εις τον εντοπισμό των εγκλημάτων σε διεθνές επίπεδο και μετά υπάρχει ο δεύτερος κύκλος που είναι πολύ σημαντικός ε, για να μετρήσει κανείς τη διαφθορά. Υπάρχουν ε, οι διαδικασίες ε, αυτοαξιολογήσεως και συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν από τον ενεργό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων και ε, βλέπουμε ότι καταρχήν συγκεντρώνονται οι εθνικές πληροφορίες από τους αναθεωρητές και συγχρόνως προωθούμε το διάλογο μέσω επισκέψεων σε διάφορες χώρες ε, με τη διοργάνωση κοινών συνεδριάσεων όπου οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ενθαρρύνονται να συμμετέχουν για να συμβάλλουν στη συζήτηση κατά τις διαβουλεύσεις με τους αναθεωρητές με στόχο να αναθεωρηθούν οι διατάξεις σχετικά με την ποινικοποίηση και την διεθνή συνεργασία. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν της αξιολογήσεως του αποτελέσματος της διαφθοράς και των εφαρμοστικών μέτρων βασίζεται σε μία αξιολόγηση ομοτήμων και μία ε, διαδικασία παράλληλη ε, διαβουλεύσεων μεταξύ της εξεταζομένης χώρας και των εξεταστών κατά τρόπον ώστε να μπορεί κανείς να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ε, και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εναντίον της διαφοράς στην εξεταζόμενη χώρα Είμαστε τώρα στον τρίτο χρόνο της αναθεώρησης. Έχουμε συγκεντρώσει ε, πληροφορίες σχετικά με, τους, ε, με τα δύο πρώτα χρόνια ε, για τα μέτρα ποινικοποιήσεως και αντιμετωπίσεως της διαφθοράς και τα πρώτα αποτελέσματα αναφέρονται τα ίδια θέματα που ανέφερα ήδη. Δηλαδή, καταρχήν διαπιστώσαμε και εμείς ότι στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη που έχουμε εξετάσει μέχρι στιγμής υπάρχει κάποια συνέπεια μεταξύ την εσωτερήκευση ορισμένων αδικημάτων ε, δωροδοκίας στην εθνική νομοθεσία νομοθεσία εις ε, το whistleblowing δηλαδή εις ε, την υπόδειξη ε, υπετίων και εις την συστηματική συγκέντρωση πληροφοριών ε, για την διεθνή ε, συνεργασία και για να δούμε πώς η ε, διεθνής αμοιβαία αρρωγή εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε συστηματικά να συγκεντρώσουμε τα αναγκαία στοιχεία και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αιτήσει οι οποίες μας έχουν υποβληθεί και σε πρακτικά θέματα που αναφέρονται σε διεθνή συνεργασία. Ένα άλλο θέμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, στη συνέχεια μετά από τις αναθεωρήσεις αυτές είναι το είδος και η ανάγκη τεχνικής βοηθείας που χρειάζεται και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για την ε, επιτυχή έκβαση της ε, αναθεώρησης ότι δηλαδή οι περισσότεροι που έχουν εντοπιστεί χρειάζονται τεχνική βοήθεια και ε, βοήθεια για την κατάρτιση προγραμμάτων ε, δράσης για την εφαρμογή της ε, διαδικασίας εφαρμογής των προγραμμάτων εναντίον της διαφθοράς. Ξέρω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος μου και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο δεύτερο επίπεδο της αξιολογήσεως της μετρήσεως της διαφθοράς πέραν του θεσμικού επίπεδου της αναθεώρησης της διαφοράς στις εξεταζόμενες χώρες. Πρόκειται για το επιστημονικό επίπεδο και ε, τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για να καταπολεμήσει τη διαφθορά στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και βεβαίως το σημείο κίνησής μας είναι ότι δεν υπάρχει μόνο μία πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την διαφθορά αλλά και διαφορετικές μεθοδολογίες η επιστημονική ανάλυση την οποία χρησιμοποιεί ο οργανισμός μας δεν βασίζεται εις, ε, ε, εις δείκτες αλλά σε διαφορετικές ποιοτικέ προσεγγίσεις δηλαδή αξιολογήσεις από ε, εμπειρογνώμονες ε, και ε, συμμετοχή σε ένα δίκτυ βασίζονται δε σε διαφορετικές προσεγγίσεις και οι πληροφορίες ε, εξασφαλίζουν ότι θα συμβάλλουν πολλές ε, ε, πηγές, τα δικαστήρια, οργανισμοί καταπολέμησης της διαφθοράς και μετά τη συγκέντρωση των πληροφοριών γίνεται μία ε, αξιολόγηση κατά τρόπον ώστε να βασιστούμε στις ε, άμεσες ε, εμπειρίες των διαφόρων εμπλεκομένων και έτσι ε, υπάρχει μία μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται από την ε, UNDC και αναφέρεται εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οτιδήποτε ερωτήματα έχετε να μου κάνετε. Προς το παρόν θέλω να σας πω ότι και από πλευράς μεθοδολογικής από σκοπιά ε, επιστημονική αλλά και στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου του μηχανισμού αναθεώρησης η βασική και ε, ουσιαστική αρχή την οποία εφαρμόζουμε είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα κατατάξεως χωρών. Ο πιο βασικός στόχος είναι ε, ο μηχανισμός ε, αξιολογήσεως που δεν βασίζεται σε κατάταξη αναλόγως ε, του αντιληπτού βαθμού διαφθοράς αλλά εντοπισμού των ελλείψεων και της επιλύσεώς τους μέσω τεχνικών μέσων και βοηθείας εάν δεν υπάρχει δυνατότητα εντοπίως να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Ή σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε. Ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση και δίνω τον λόγο στον εισηγητή κύριο Γιακολίνο. Ε, είχαμε λοιπόν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις ε, και είχαμε και έχουμε και την εισήγηση που θα συνταχθεί με την βοήθεια όλων των πολιτικών ομάδων και με όλα αυτά βέβαια που ακούσαμε σήμερα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις απόψεις μου είναι σαφές ε, ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια σειρά δικτών για να μπορούμε να μετρήσουμε την έκταση της ε, διαφθοράς και είναι και σαφές ότι ποικίλουν τα κριτήρια από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Επίσης ε, είναι σαφές ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει τεχνική βοήθεια όσον αφορά τις ε, οργανώσεις που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ. Και αυτό για να μπορέσουμε να ελέγξουμε ένα φαινόμενο το οποίο ε, και μόνοι σας είπατε ότι αυτή τη στιγμή επεκτείνεται. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις ξεκινώντας από το εξής. επειδή ελέγχθησαν κάποια πράγματα, θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσουμε πώς ακριβώς φτάσαμε στο να έχουμε ένα ΑΕΠ που αφαιρείται από τον πλούτο της οικονομίας μιας χώρας λόγω της ε, διαφθοράς η οποία έχει παρισφρήσει σε όλους τους κλάδους της ε, δημόσιας διοίκησης. Επίσης, μήπως μπορείτε να μας πείτε ε, και τι συμβαίνει με τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα σε επίπεδο ιδιωτών. Έγινε αναφορά στην Κίνα ε, τι ακριβώς συμβαίνει στην Κίνα σε σχέση με την ενημέρωση από τη χώρα αυτή και νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, επίσης, τελειώντας, θέλω να πω σχετικά με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες. Ε, αναφέρομαι στη χρηματοδότηση των κομμάτων και της πολιτικής νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξουμε στην εισήγησή μας και αυτό διότι θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια σωστή προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά που σας ανέφερα και αυτά θεωρώ ότι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην ε, τελική έκθεση. Τέλος, όσον αφορά το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο ε, πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο όσον αφορά σε αυτό το φαινόμενο που αναμφίβολα υπάρχει στα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιακολίνο εκ μέρους της, ε, των φιλευθέων. Ο κύριος Νιούτον Ντάν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Και έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά και τους τρεις ε, ομιλητές, ε, γιατί μιλήσατε κατ' ουσίαν για το ίδιο θέμα, αλλά από, διαφορετική, από διαφορετικό πρίσμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα απόλυτο κριτήριο για το τι είναι η διαφθορά και τι όχι. Νομίζω πως όχι. Όλα σχετικά είναι. Και από χώρε όπως ε, η Κίνα, ε, τι είδους αντιδράσεις ε, έχετε. Βλέπουμε ότι οι τράπεζες ε, της Κίνας είναι στο κάτω μέρος του καταλόγου. Το να λέμε ότι οι τράπεζες της Κίνας είναι ανοιχτές, αυτό είναι αστείο τουλάχιστον με τα δικά μας κριτήρια. Όπως και πολλά άλλα θέματα στη ζωή, όλα είναι υποκειμενικά. Και μία άλλη ερώτηση. Από την δική σας την εμπειρία, τι είδου ε, αλλαγές ε, πρέπει να γίνουν ε, σε μία χώρα. Γιατί φαίνεται ότι η Ευρώπη είναι χειρότερη στα μάτια των πολιτών. Όχι διότι δεν υπάρχουν οι νόμοι, συνεχώς θεσπίζουμε νόμους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι είδου αλλαγές έχουν γίνει για τη διαφθορά από χρονιά σε χρονιά. Αυτά, από ό,τι φαίνεται, γίνονται κάτω από τα μάτια μας, αλλά μοιάζει να μην τα βλέπουμε εκ μέρου του ΕΛΚΟ, κύριος, η κυρία Ματιό, με Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους τρεις ομιλητές. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις. Θα αναφερθώ σε εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας και του UNODC. Μας δώσατε πολλούς δείκτες, ε, αλλά οι οργανισμοί σας ε, ουσιαστικά πρέπει να κάνουν και κάτι ακόμα. Δηλαδή, εφόσον έχετε εντοπίσει ένα λόγο διαφθοράς, τι συμβαίνει στη συνέχεια, τι κάνετε. Τι κάνουν οι δικοί σας οργανισμοί, δηλαδή ε, θέτετε κάποιο εμπόδιο σε αυτή τη διαφθορά στις καταβολές ε, γιατί εμείς μπορεί να έχουμε ε, κάποια αρμοδιότητα σε σχέση με την ομοθεσία, όμως εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι ε, πρακτικό, το κάνετε. Και κατόπιν ε, να αναφερθώ, κυρία Μιτμάιερ, στη δική σας ομιλία. Τα είπατε πάρα πολύ γρήγορα, ήταν πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα. Εγώ ήμουν διακοπές στην Ασία, όχι στην Κίνα, αυτό το καλοκαίρι. Και ε, μπορώ να σας πω, ναι, μεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφθορά, αλλά στην Ασία είναι τρομερή κατάσταση. Σε αυτές τις δύο χώρες... Ε, που πήγα εγώ ήταν τεράστια διαφθορά. Μία γυναίκα έπρεπε να κάνει και σαρική και έπρεπε να καταβάλει φακελάκι κατά κάποιο τρόπο, έπρεπε να περιμένει και αν ε, δεν ε, καταβάλλεται ε, αυτό το φακελάκι δεν μπορεί να γίνει τίποτα και επίσης να περάσει κανείς τα σύνορα έπρεπε ε, να πληρώσει ένα ε, κατά κάποιο τρόπο και καθημερινά σχεδόν συνεβαίνε αλλά σχεδόν για να περάσει ένας να διασχίσει κάποιος από τον ένα δρόμο στον άλλο επερβάλλω αλλά κάτι τέτοιο συνέβαινε στις δύο χώρες που πήγα εγώ πραγματικά μπορώ να σας πω ότι ήταν φιαλτική κατάσταση για τους πολίτες ε, καθώς και το επίπεδο ζωής τους είναι τρομακτικό. Και πέρα ε, από το ότι πρέπει να πληρώνουν ε, αυτά τα ποσά πρέπει να βρίσκουν και τρόπους να εξασφαλίσουν αυτά τα ποσά. Δεν ξέρω πώς επιβιώνουν λοιπόν. Έτσι λοιπόν σας ευχαριστώ που προσπαθείτε εσείς να θεσπίσετε κάποιους δείκτες για κάποιους τρόπους ανάσχεσης. Σας ευχαριστώ. Κύριο Σμιτ. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, καθυστέρησα σήμερα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γνωρίζω ότι όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κομμάτων υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη χώρα μου τη Σουηδία το οποίο όμως εμείς το εξετάζουμε. Βέβαια εδώ οι κύριοι που μίλησαν έφυγαν. Εγώ να σας πω πάντως ότι προοδεύουμε, προχωράμε στο θέμα αυτό. Ε, και όλα αυτά δείχνουν ότι δείχνουν και τον τρόπο που ψηφίζουμε. Τέλο πάντων, εμεί στη Σουηδία κάπω το παλεύουμε το θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποιε βόρειε χώρες ε, που υποτίθεται ότι είναι καλύτερες. Και ερωτώ, γιατί υποτίθεται ή γιατί εμφανίζονται ως καλύτερες λόγω του κλίματος, λόγω του κράτους πρόνοιας, λόγω του φορολογικού συστήματος. Ε, εσείς γελάτε, δεν ξέρω, ίσως αυτά να μην ισχύουν στη Δανία, αλλά νομίζω ότι είναι ε, ενδιαφέρουσα αυτές οι ερωτήσεις. Μήπως είναι λάθος η άποψη που επικρατεί. Γιατί πρέπει να σας πω ότι και εμείς ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε τεράστια σκάνδαλα. Αλλά δηλαδή μην πιστεύετε ότι είμαστε άγγελοι. Και μία άλλη ερώτηση. Διότι και ο Μπιλ αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα υπάρχει πράγματι άμεση σχέση ανάμεσα στη δημοκρατική ανοιχτή κοινωνία και, μια λιγότερο δημοκρατική. Εγώ έχω δει κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι ε, άσχετα τα δύο πράγματα μεταξύ τους. Μερικές χώρες, ακόμα και ανοιχτές δημοκρατικές ε, κοινωνίες μπορούν ε, να είναι λιγότερο διεφθαρμένες. Πάντως σας ευχαριστούμε όλα αυτά που είπατε είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά καταλήγουμε στο ότι λίγο πολύ εδώ, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αυτό το χώρο, είμαστε ε, όλοι διεφθαρμένοι. Η κυρία Γκόμες. Η κυρία Γκόμες. Πρέπει να σας πω στην Βερονίκ Μαρτιό ότι δεν χρειάζεται να πάμε στην Ασία για να δούμε τα, ε, τη διαφθόρα αλλά ε, στην Πορτογαλία τώρα με την παρέμβαση της Τρόικα και βλέπουμε ε, γέρους που πάσχουν από καρκίνο και από χρόνιες ασθενείες και που δεν πάνε στο νοσοκομείο γιατί δεν έχουν χρήματα και δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους που τους επιβάλλουν για την υγειονομική περίθαλψη ή δεν έχουν χρήματα για τη μεταφορά τους. Θέλω να ρωτήσω τους τελευταίους ομιλητές. Ε, Ε, κοιτάξτε, το θέμα της ε, έκθεσης ε, δεν είναι αυτό το χειρότερο, διότι το πρόβλημα που υπάρχει είναι να αντιμετωπίσουμε την ατιμορρησία σε σχέση με τη διαφθορά και, την και το οργανωμένο έγκλημα. Και βλέπουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη δικαστική εξουσία, είτε διότι δεν έχει τα μέσα, είτε διότι και αυτή είναι διεφθαρμένη. και το σημαντικότερο, το πιο αποτρεπτικό στοιχείο είναι η έκθεση. Έτσι λοιπόν ρωτώ τι κάνουν οι οργανώσεις για να εκθέσουν τους διεφθαρμένους και για να αποκαλύψουν ότι η φορολογική παράδειση σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ακριβώς οι μαύρες εκείνες τρύπες που επιτρέπουν να υπάρχει αυτή η διαφθορά και η χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος. Τι κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα, ας πούμε, για να εκθέσει την Delaware την τον Τέλεγορ σαν ένα μεγάλο φορολογικό παράδεισο κοντά στην Ουάσιγκτον ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ έχουμε φορολογικούς ε, παραδείσους ε, που είναι και νόμιμοι. Να σας πω το εξή. Η δική μου η χώρα και η παρέμβαση της ε, Τρόικα διαπίστωσε ότι μόνο μία από τις 20 εταιρείε ε, που έχουν εισαχθεί ε, στο χρηματιστήριο έχουν ε, τους, ε, τις έντρες τους ε, εκτός Πορτογαλίας. Μόνο μία έχει έντρα στην Πορτογαλία και ξέρετε γιατί το κάνω αυτό για να πλέουν λιγότερους φόρους. Να πλέουν ας πούμε στην Ολλανδία που είναι χαμηλότερη η φορολογία το εντέταρτον τέταρτον αυτής που ισχύει στην Πορτογαλία και ξέρετε κάτι αυτό θεωρείται νόμιμο αλλά με συγχωρείτε αυτό είναι παράνομο, είναι παντελώς παράδοξο. Για να μην αναφέρω και όλες τις άλλες συναλλαγές ε, που γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο με διεφθαρμένο τρόπο. Η έκθεση λοιπόν, η αποκάλυψη. Ε, πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωσης ε, παίζουν καθοριστικό ρόλο, αλλά και οργανώσεις σαν τη δικιά σας μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για να βοηθήσουν τα μέσα ενημέρωσης να αποκαλύψουν όλα αυτά εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι στην Επιτροπή μας προσπαθούμε να το κάνουμε και μόνοι μας βέβαια. Ε, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε και κατά την άποψή μου ε, η αποκάλυψη ε, αυτών των ανθρώπων και των οργανισμών είναι το σημαντικότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι αρκετά σαφές το πλαίσιο μέσα στο οποίο τέθησαν οι ερωτήσεις. Δηλαδή, οι ερωτώντες όχι μόνο δήλωσαν ότι τους άρεσαν πάρα πολύ ομιλίες, αλλά εγώ πιστεύω ότι και εσείς ε, είναι απαραίτητο να δίνετε ε, πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, ίσως να μπούμε ακόμα περισσότερο σε λεπτομέρειες. Και ίσως αυτό θα ήταν και χρήσιμο για τις ε, εργασίες της Επιτροπής. Να γνωρίζουμε λοιπόν ποιες είναι οι χώρες εκείνες και κυρίως ε, σε ποιο πλαίσιο και με ποια μέθοδο μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Ε, προηγουμένως ε, έγινε λόγος από τον κύριο Νιούτον Ντάν ε, για τις ασιατικές χώρες και για την Κίνα. Πρόσφατα το καλοκαίρι πήγαμε στη Σερβία και είχαμε εκεί τον τρόπο να θέσουμε το δάκτυλο στον τύπο των ήλων στην διαδεδομένη ε, διαφθορά ας πούμε καταρχήν στην αστυνομία γιατί η αστυνομική κερδίζουν πάρα πολύ λίγα χρήματα, είναι χαμηλόμιστη. Και πολύ συχνά όταν ε, ε, επιβάλλουν ένα πρόστιμο ο πολίτης ξέρει ότι αν προσφέρει στον αστυνομικό το ίμιση του προστίμου, του ποσοποντιστοιχεί στο πρόστιμο, ο αστυνομικός δισκίζει βάζει τη, τα μισά στην τσέπη και τελειώνει η ιστορία. Αυτό ε, μας παρουσιάστηκε σαν κάτι το φυσιολογικό. Δηλαδή ένα στοιχείο που βοηθάει κάποιους να επιβιώσουν, απ' την άλλη όμως ε, επιβάλλει μια στάση που μοιάζει να είναι φυσιολογική και το ίδιο και όταν ε, ήρθαμε σε συζητήσεις ε, με τα διάφορα στελέχη της διοίκησης. Αυτό εμείς το εντοπίσαμε, αλλά δεν νομίζω ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Ακόμα και ο κύριος Σμίτ είπε ότι και εμείς στη Σουηδία έχουμε μεγάλα προβλήματα δεν νομίζω ότι είναι κανείς ε, αλόβητος. Ε, όλοι έχουν προσβληθεί από την διαφθορά. Αλλιώς δεν θα μιλάγαμε σήμερα για το θέμα αυτό. Ή αλλιώς η Επίτροπος κυρία Μάλστρομ ε, δεν θα μιλούσε για το θέμα αυτό που κατά τη δική μου άποψη το είπε μάλιστα και πάρα πολύ συγκρατημένα γιατί η Επίτροπος μίλησε για 120 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο που λίγα μου μοιάζουν γιατί με βάση τα στοιχεία των ελεγκτικών συναντρίων ε, το Ιταλικό και το Ευρωπαϊκό αυτά τα 120 στα 120 δις, από τα 120 δις, τα μισά, τα 60 αφορούν την Ιταλία. Και η κυρία Μίτερμα αναφέρθηκε στην ταξινόμηση των χωρών. Η τελευταία είναι η Βουλγαρία. Τρίτη από το τέλος είναι η Ιταλία. Μιλάμε τώρα για χώρες ε, οι οποίες είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επίπεδο αποδοχής και η σύγκριση που γίνεται εγώ νομίζω ότι είναι απαράδεκτο Οφείλουμε λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι όχι να γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο αρχής, αλλά ε, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, να μην τα μπερδεύουμε, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να τα αναφέρουμε τα κράτη αυτά, γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε γύρω-γύρω από τα προβλήματα, χωρίς να βάζουμε, όπως είπα, το δάχτυλο στον τύπο των νερών, καμία χώρα δεν θα καταλάβει ή δεν θα θεωρήσει ότι φύγεται. Εμείς λοιπόν αυτή τη δουλειά την κάνουμε με αίσθημα ευθύνη και ξεκινάμε από την παραδοχή ότι εάν στα δικά μας τα κράτη υπάρχουν προβλήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το να μην τα αντιμετωπίζουμε αυτό δεν σημαίνει ότι προσφέρουμε υπηρεσίες ε, στη χώρα μας. Ε, το να επισημάνει κανείς κάτι δεν σημαίνει ότι δυσφημεί κανείς τη χώρα του. Θα πρέπει να δείξουμε τα πράγματα με ειλικρινή τρόπο. Γιατί αν προσπαθούμε κάπως ε, να τα συγκαλύψουμε γιατί αλλιώς ενδεχομένως ε, να προκύψει πρόβλημα στη χώρα, η χώρα να γίνει αντικείμενο συζητήσεων ανά τον κόσμο. Αυτό είναι λάθος. Ε, λάθος υπηρεσίες προσφέρουμε στους πολίτες μας, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση. Αν λοιπόν συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε αυτήν την επιπολαιότητα, φοβάμαι ότι ε, τα πράγματα ε, θα φτάσουν στο σημείο μηδέν. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ στους ε, προσκεκλημένους μας και να τους πω θέλω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ήθελα να αναφέρετε, να κατονομάσετε τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά βέβαια αυτό σας το ζητώ με απόλυτη σύνεση γιατί εδώ η δουλειά που κάνουμε δεν θα πρέπει να είναι δουλειά βιτρίνας. Εμείς έχουμε βάλει στόχους, ε, θέλουμε να προχωρήσουμε με βάση τους στόχους που έχουμε θέσει και μόνοι μας πολλές φορές έχουμε μιλήσει για δυσκολίες που υπάρχουν. Μιλήσαμε χτες ε, για το πόσο δύσκολο είναι να περάσει κανείς ε, στην εναρμόνιση των ε, διοικητικών ε, δικαστικών συστημάτων. Αλλά αν δεν αρχίσουμε σιγά σιγά βήμα προς βήμα να, να κοιτάμε και τα του οίκου μας και όταν μιλάω για τα του οίκου μας αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θα ε, κάνουμε πολλά αλλά δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Για να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Εγώ πιστεύω αυτή η Επιτροπή όχι μόνο θέλει να είναι αποτελεσματική αλλά έχουμε, χρειαζόμαστε να μας ε, πείτε ποιες είναι οι χώρες σε εκείνη την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πρωταθλήτριες ε, στην ε, διαφθορά. Ε, δεν θέλω να στυλιτεύσω μια χώρα περισσότερο από άλλη, αλλά είναι σημαντικό για να ξέρουμε από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, τι είδου λάθη έχουν γίνει, ποια είναι τα επιπόλαια στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Το πρόβλημα είναι τεχνικής φύσεως αλλά και πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ ε, να ε, μπείτε λιγάκι σε βάθος ε, στις εισηγήσεις σας και θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την συνάδελφο από την Ιταλία. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα θέματα και στις ερωτήσεις που τέθηκαν μέσα σε κάποια λεπτά. Όλα τα θέματα που τέθηκαν είναι θέματα για τα οποία εγώ αγωνίζομαι καθημερινά. Θυμάμαι το ρόλο που διαδραμάτισα ως εκπρόσωπος ενός οργανισμού που πήγα σε μια χώρα και να σας ξεκαθαρίσω το εξή. Όταν πρόκειται για τη διαφθορά, η Παγκόσμια Τράπεζα δεν μπορεί να θέσει αυτό το θέμα με τη χώρα. Η χώρα καλεί ρωτήστε την κυβέρνησή σας. Γιατί εμάς μας δικούν εκπρόσωποι από κάθε κυβέρνηση στον κόσμο. Μπορούμε να μιλήσουμε για τη διαφθορά, είναι παντού στα εγγραφά μας αυτό το θέμα, αλλά εγώ δεν μπορώ να απομονώσω αυτό στο πιο σημαντικό ζήτημα. Σε μία σχέση μπορώ να θέσω ότι υπάρχει δυνατότητα προσυζήτηση, αλλά θα πρέπει να προσκληθώ να πάω εκεί και να συζητήσω συγκεκριμένα για πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και για να φερθώ στο είπε η κυρία Ματιέ, τι κάνουμε να ε, σταματούμε το δανεισμό, ποια είναι η στρατηγική μας, αν ε, δούμε ότι μια χώρα δεν συμπεριφέρεται με ικανοποιητικό τρόπο. Πάντοτε δίνουμε τη βοήθεια γιατί θυμηθείτε το στόχο της Παγκοσμία Τράπεζας που είναι διαφορετικός. Εμείς θέλουμε να προσπαθήσουμε να εξελίψουμε τη φτώχεια. Έτσι λοιπόν, ε, περίπου πριν πέντε χρόνια, Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα κάνουμε. Κάποιοι από εμά θεώρησαν ότι έπρεπε να σταματήσουμε να παρέχουμε πόρου ε, σε χώρε και κυβερνήσει ε, που δεν του χρησιμοποιούσαν με τον κατάλληλο τρόπο και άλλοι θεώρησαν όχι, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον ε, να συνεργαστούμε με ένα τμήμα τη χώρας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι γιατί διαφορετικά αυτοί που θα πληρώσουν το τίμημα θα είναι οι πιο φτωχοί. Όμως θυμηθείτε ότι συνεργαζόμαστε με χώρες που δεν ε, είναι το είδο τη Ευρώπη που έχετε, το τη χώρα μα που έχετε στην Ευρώπη. Πρόκειται για διαφορετική πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, οι κυβερνήσει ε, όλων των χωρών στον κόσμο εκπροσωπούνται στην Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτή είναι. Και εγώ διαβάζω αυτό σημάδι των καιρών για το επίπεδο της πολιτικής βούλησης εγώ ως τεχνοκράτης ε, τώρα στο ιστορικό της Παγκόσμιας Τράπεζας έχω κάποια επιλογή και να είμαι πολύ συγκεκριμένη. Αν ε, υπάρχει διαφθορά σε μια χώρα και πιστέψτε με, οι χώρες ε, όπου ταξιδεύω εγώ είναι σαν τις χώρες όπου είδατε αυτά που είδατε. Τι κάνουμε. αν ε, βλέπουμε, ε, βλέπουμε μία διαφορά στο επίπεδο της διαφθοράς ε, σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε κάποια αποδεικτικά στοιχεία και έχουμε εμπειρία και συστήνουμε στις χώρες τι θα κάνουν. Διαφάνεια, ε, έκθεση και πρέπει να συνοδεύεται και με επιβολή του νόμου. Γιατί μόνο η έκθεση, χωρί να υπάρχει κάποια συνέπεια, μόνο η καταγγελία χωρί να υπάρχει κάποια συνέπεια, δεν έχει νόημα. Έτσι λοιπόν τα δύο αυτά μαζί είναι σημαντικά. Αν σκεφτούμε τη διαφθορά που είναι ενδημική στο δημόσιο τομέα, ένα άλλο στοιχείο που βρήκαμε και είναι πολύ σημαντικό είναι η λογοδοσία. Και τι εννοώ να έχουμε ένα δημόσιο τομέα που ουσιαστικά λειτουργεί χρησιμοποιώντας αξιοκρατικά πρότυπα. Είναι διαφανής στον χειρισμό των πάντων, στο πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι, οι χρηματοοικονομικοί πόροι, οι ανθρώπινοι πόροι και οι διαθέσιμες πληροφορίε. Όταν ε, λοιπόν καθόμουν στο τραπέζι με τις κυβερνήσεις ε, και μόλις ε, επέστρεψα από το Κάιρο, και εκεί συνεργάστηκα με διάφορους εκπροσώπους όλων των χωρών της Μέσης Ανατολής, αυτό τους λέμε. Ελέγξτε αν υπάρχει πολιτική δέσμευση για να γίνει τι και πόσο μακριά και αν μπορείτε να το υποστηρίξετε και κατόπιν. Να δούμε. Θέλετε να επικεντρωθούμε στο να βελτιώσουμε στο πώς χειρίζεστε τους ανθρώπινους πόρους, ε, τους υπαλλήλους σας ή αν θέλουμε να επικεντρωθούμε στις δημοσίες συμβάσεις και να καταστήσουμε τη διαδικασία πιο διαφανή και να υπάρχουν και συνέπειες αν ανακαλύψουμε ότι στη διαδικασία υπάρχουν παρατυπίες. Γιατί απλώς ε, το να διαθέτουμε κάποιες πληροφορίες χωρίς να υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, κάτι τέτοιο δεν βοηθά. Και εδώ βλέπετε τη διαφορά. Μια χώρα στην Ευρώπη που επηρεά... οι χώρες στην Ευρώπη που επηρεάζονται λιγότερο από τέτοιες συμπεριφορές είναι οι χώρες όπου εφαρμόζονται οι νόμοι, που εφαρμόζονται αυτές οι αρχές. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρον με κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Global Integrity και ε, ερευνά τι και να υπάρχουν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας ε, στις χώρες. Σε χώρες όπως η Ουγγάντα, όπου έχουν ένα πολύ καλό ποσοστό σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, έχουν όμως το πιο μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δηλαδή υπάρχουν νόμοι, αλλά κανείς δεν τις εφαρμόζει. Ποιο είναι το νόημα λοιπόν. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο και θα καταλάβετε γιατί η δουλειά μας ε, δεν είναι τόσο απλή. Ένα στοιχείο ε, είναι το πώς ε, θα ε, διαχωρίσουμε τις χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος διαφοράς από αυτές που υπάρχει μικρότερος. Είναι το θέμα της ε, ικανότητας. Ε, δηλαδή, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίε πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός ικανότητας δυναμικής στη χώρα αυτή. Και αυτό είναι σημαντικό. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά το θέμα αυτό όταν ε, σχεδιάζουμε ένα, μία δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση τη διαφθορά, επιτρέπουμε στη χώρα να μετρήσει τη διαφορά, να, κατανοήσει, που είναι τα προβλήματα, να οικοδομήσει αυτέ τι ικανότητε και να του δώσουμε ένα εργαλείο σχετικά με τη λογοδοσία, την πρόσβαση την πληροφορία και τη διαφάνεια. Και κατόπιν, ε, μεσοπρόθεσμα, υπάρχει εφαρμογή. και αν σκεφτούμε κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν, γιατί τώρα βλέπουμε τόσο πολύ περισσότερη διαφθορά στην Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι φαινόμενα που πάντοτε ήταν παρόντα και πριν 20 χρόνια, όταν εγώ πήγαινα σχολείο, με για το λίπος, το λάδι που είναι απαραίτητο για να κινείται η οικονομία, θα το θυμάστε. Δηλαδή ήταν απαραίτητο να έχουμε επιτυχή επιχειρηματικότητα. Έτσι το παρουσίαζαν 20 χρόνια πριν, 20 χρόνια μετά. Διαφέρουν τα πράγματα και συζητούμε πολύ περισσότερο για αυτό το θέμα. Επομένως υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία. Και θέλω να επανέλθω στο θέμα της ε, έκθεσης, της αποκάλυψης. Ε, ναι, για να καταπολεμηθεί η ατιμορρυσία. αλλά μόνο όταν υπάρχει εφαρμογή της νομοθεσίας. Στην Παγκόσμια Τραπέζα εγώ έχω πάρα πολύ υλικό. Ευχαριστώ να σας το μοιράσω, να σας ε, δώσω πληροφορίες για το που βρίσκονται τα διάφορα δεδομένα. Επίσης, ε, προσπαθούμε να δούμε πώς στη δημόσια δίκηση μιας χώρας ε, εφαρμόζεται η νομοθεσία σε σχέση με τη δημοσίευση των πληροφοριών, τι γίνεται με την προστασία της ασυλίας, με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τι γίνεται με την εφαρμογή όλων αυτών, γιατί αν δεν εφαρμόζονται αυτά τα κυρία νομοθετήματα, πραγματικά αγωνίζεσαι να έχεις ένα σύστημα που ακόμη και αν υπάρχει παρουσία κινδύνου διαφθορά, τότε θα μπορεί να απαντήσει τον κίνδυνο αυτό. Και ο κίνδυνο διαφθορά υπάρχει σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Δεν ε, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει μηδενική διαφθορά σε κάποια χώρα. Απλώ πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι χώρε έχουν συστήματα που να μπορούν να απαντήσουν σε οποιοδήποτε είδο ενδυνάμει κινδύνου. Γιατί η διαφθορά θα του λήξει και θα σκεφτούν ένα νέο τρόπο να υπάρξει μια συναλλαγή που να υπερβαίνει τον νόμο. να παρακάμπτει τον νόμο. Τώρα για τη συγκεκριμένη ερώτηση που τέθηκε σχετικά με τη διαφθορά δύο ιδιωτικών υπηρεσιών και για τον ορισμό της διαφθοράς. Όταν σκεφτόμαστε τη διαφθορά και θα επανέλθω στο σχόλια του κ. Γιακολίνο, μιλάμε για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος για ίδιο Δηλαδή μια τυπολογία διαφθοράς που εμπλέκει κάποιον που είναι δημόσιος υπάλληλος και κάποιον που είναι εκτός της υπηρεσίας. Πολύ καλά αναφερθήκατε στη διαφθορά που υπάρχει μεταξύ δύο ιδιωτικών οντοτήτων που πραγματικά μπορούν να στερευλώσουν την οικονομία μιας χώρας. Πρόσφατα αρχίσαμε να σκεφτόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να σταματήσουν αυτό το φαινόμενο. Φυσικά και η αρχή που αναφέρα πριν θα εφαρμόζεται εκεί, αλλά έχουμε πολύ λιγότερα παραδείγματα. Πρόσβαση στις πληροφορίες, λογοδοσία, όλα αυτά ισχύουν, αλλά... Συγκεκριμένα παραδείγματα έχω πολλά σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς μίσους της διαφθοράς ε, μεταξύ ενός δημοσίου υπαλλήλου και ενός ιδιωτικού υπαλλήλου. Όμως όταν έχουμε δύο ιδιωτικού φορείς υπάρχουν πολύ λιγότερα παραδείγματα. Και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία γιατί είναι δύσκολο να βρούμε και τις περιπτώσεις διαφθοράς εκεί. Και επίσης για το σύνδεσμο μεταξύ διαφθοράς και δημοκρατίας, ε, ερώτηση που τέθηκε από κάποιον, αυτό ο σύνδεσμος είναι εντελώς ασαφής. Και ευχαρίστω ε, να πω δύο λόγια γι' αυτό. Το ελεκτικό συνέδριο Ε, διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε περί μεταρρύθμιση σε μία χώρα, όχι μόνο πρέπει να ενδυναμώσουμε τις, ε, τη δημόσια διοίκηση, αλλά πρέπει να ενδυναμώσουμε και τους οργανισμούς εποπτείας, τους φορείς εποπτείας. Και τώρα ένα θεμελιώδες ερώτημα που έθεσε η Πρόεδρος αν πρέπει να δακτυλοδείξουμε κάποια χώρα, υπάρχουν τα δεδομένα. Εδώ έχουμε 45 δείκτες διαθέσιμους για οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Ήδη τις διαθέσαμε στην Κομισιόν, τους δείκτες αυτούς για την έκθεση. Είναι δημόσια όλα αυτά, μπορείτε να το ελέγξετε. Εγώ δεν έχω ε, διαλέξει κάποια ευρωπαϊκή χώρα, έχω διαλέξει το Περού. Μπορείτε να δείτε του δείκτε θα καταλάβετε σε ποιο βαθμό είναι τα προβλήματα και αυτό μπορεί να σας βοηθήσει. Και όχι επειδή δεν θέλω να πάρω θέση, αλλά υπάρχουν τόσε πολλέ μορφέ διαφθορά που ίσως σε μια χώρα μπορεί να έχετε, προσπαθ... να έχετε κατορθώσει να καταπολεμήσετε τη διαφθορά παραδείγματο χάρη στον τομέα της υγείας ε, σε άλλου τομεί, αλλά όχι στι δημόσιε συμβάσει. Παραδείγματο χάρη έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε πού είναι τα καλά παραδείγματα και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούν αυτά τα παραδείγματα να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν καλά παραδείγματα και ευχαρίστω να μοιραστώ μαζί σας όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μητερμαϊρ, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. σχετικά με το θέμα του τι αλλαγές επιφέρει σε μία χώρα η διαφθορά αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε μια χώρα για να αλλάξει η ατμόσφαιρα και το θέμα της διαφθοράς είναι κάποια σαφή ένδειξη από την κορυφή ότι το κράτος αντιτίθεται στην διαφθορά πρέπει να λέγεται σαφώς και ευθέως και να περνάει και παντού προς τα κάτω. Ε, επίσης ε, όσον αφορά ε, τους ελεγκτικούς οργανισμούς χρειάζεται πέραν αυτού ένας οργανισμός για την διαφθορά και υποχρεωτικούς ε, κανόνες και νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων και με ε, τις ποινές ε, για τους διεφθαρμένους δημοσίους λειτουργούς. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε στην Κίνα, η δεύτερη ερώτηση, όλες οι οργανώσεις στον κόσμο μπορούν να είναι υπόλογες μόνο αν έχουμε επαρκή πληροφόρηση. Οπότε στα οικονομικά θέματα και στις επιχειρήσεις θα πρέπει οι εταιρείε να μας πούν τι πρόγραμμα έχουν εναντίον της διαφθοράς, τι ε, είναι οι πρακτικές που εφαρμόζουν για τις συναλλαγές με τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό, όπου έχουμε γενικές αρχές περιλαμβάνουμε και τις ε, τράπεζες και τις εταιρείες της Κίνας ε, που κινητοποιούνται διεθνώς και ζητούμε να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται ε, με τις αρχές μας και αυτό αποβλέπει στο να έχουμε ε, ίσες συνθήκες για όλους διότι διαφορετικά δεν θα ε, επιτύχει το σύστημα. Βέβαια ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, υπάρχει ήδη ε, υποχρεωτικός έλεγχος ο οποίος είναι ένα μεγάλο προσόν και ελπίζουμε ότι θα έχουμε επιτύχει τους ίδιους κανόνες και είμαι πολύ ευτυχής και μπορώ να σας ενημερώσω ότι πριν από μισή ώρα ε, ψηφίσαμε τους κανόνες αυτούς και οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς της ε, εξορυκτικές βιομηχανίες για πετρέλαιο και ε, αέριο και είμαστε ε, πιο κοντά στην διαδικασία συναπόφασης να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για τις ε, ε, ε, εταιρείε οι οποίες κινητοποιούνται στο εξωτερικό και το επιζητούμε και στις τηλεπικοινωνίες και στον τραπεζικό τομέα. Η υιοθέτηση λοιπόν αυτών των κανόνων στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας προωθήσει. Ελπίζουμε ότι δεν θα αναποδυναμωθεί από το Συμβούλιο και ότι θα ενισχυθούν οι ε, κανόνες ενημέρωσης ε, για όλες τις βαθμίδες. Επίσης, ε, αν θέλετε περισσότερες προφορίες σχετικά με την έρευνά μας και τις απόψεις μας, μπορείτε να μας στείλετε μία, ένα μήνυμα ηλεκτρονικό. Ο, ο κύριος Χρυσικός. Ευχαριστώ. Πολλά από τα ερωτήματα είναι πολύ σημαντικά διότι σήμερα και κάθε μέρα προσπαθούμε ε, να βρούμε τις σωστές λύσεις και ε, ξεκινώ με το θέμα της διαφθοράς ε, μεταξύ των ε, ιδιωτών που έθεσε ο κύριος Γιακολίνο. Βεβαίως είναι ένα σημαντικό θέμα. Ε, δεν είναι μόνο η διαφθορά στον δημόσιο τομέα όπου οι εταιρείε πρέπει να καταρτήσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο για να αντιμετωπίζουν τη διαφθορά και στον ιδιωτικό τομέα συμμορφωνόμενοι με τη της διεθνής συμβάσεις ε, της ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ σχετικά με τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να πατάξουμε το φαινόμενο όταν ε, διαπιστώνουμε έξαρση της διαφθοράς σε ορισμένες χώρες. Το... Ο μηχανισμός της UNCTAD δεν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει ε, ε, επαρκής ε, κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβιάσεων των κανόνων αλλά όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ανεπάρκειες πρέπει να εμπλακούμε πιο ενεργά και να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν ευθύνες των οργανισμών μας. Πρέπει δηλαδή να συνεργαστούμε με τις εθνικές αρχές κατά τρόπον ώστε ε, να επιλύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν είτε στον δικαστικό τομέα ή στον αστυνομικό ή στην εφαρμογή. Τι γίνεται για να αποκαλύψουμε ορισμένα προβλήματα και προκλήσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό που είναι βασικό καταρχήν είναι να εξασφαλίσουμε δημοσιότητα και στα πλαίσια της δημοσιότητας προσπαθούμε να διαθέσουμε και να κοινοποιήσουμε τα συμπεράσματα των ε, εξετάσεων ε, των εκθέσεων που εξετάζουν τις διάφορες χώρες ε, που εστιάζονται στις ελλείψεις, στα προβλήματα και προβαίνουν σε συστάσεις για περαιτέρω ενέργειες των κρατών αυτών. Βέβαια η δημοσιότητα θα πρέπει να συνδυάζεται με εφαρμογή μέτρων κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν τα προβλήματα. Αλλά η εφαρμογή είναι ε, αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και είμαστε στη διάθεσή τους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Όσον αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν στην νομοθεσία των κρατών ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όπως σας είπα, δεν υπάρχει μια κατάταξη και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ποιες είναι οι χώρες σε μια περιοχή που έχουν την καλύτερη ή την χειρότερη πολιτική εναντίον της διαφθοράς αλλά έχουμε τα, τις εξελεκτικές περιλήψεις οι οποίες ε, δημοσιεύονται από την Επιτροπή ε, μας κατά τρόπον ώστε να εντοπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν και την τεχνική βοήθεια που ενδέχεται να, ε, να χρειάζεται. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Σερβία, διότι άκουσα ότι ε, θα επισκεφθείτε τη Σερβία και εμείς θα το πράξουμε την επόμενη εβδομάδα. Και βασιζόμαστε στις συμπληρωματικές δράσεις μεταξύ οργανώσεων. Το δε πρωί ε, σήμερα ακούσαμε ότι υπάρχουν εκθέσεις από διάφορους ε, οργανισμούς που παρακολουθούν τις εξελίξεις και εμείς το ίδιο κάνουμε ε, γνωρίζουμε τι κάνουν και άλλες οργανώσεις και μπορούμε να προβούμε σε κοινέ ενέργειες για να δούμε παραδείγματο χάρη στη Σερβία ε, τι συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να βοηθήσουμε τις διάφορες αρχές. Πέραν αυτού, γιατί θεωρούνται ορισμένες χώρες ότι είναι καλύτερες όσον αφορά τα μέτρα κατά πολέμησης ε, της διαφθοράς. Ε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα κλίματος ή ε, παιδείας, αλλά κατ' εμέ είναι θέμα σωστής εφαρμογής των αποτελεσματικών μέτρων να υπάρχει επαρκής μηχανισμός και ε, να υπάρχει και το αντίστοιχο πλαίσιο το οποίο να λειτουργεί σωστά ε, και μέτρα ε, και κυρώσεις εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο της διαφθοράς και ποια είναι τα ε, συγκεκριμένα θέματα που επηρεάζουν τη διαφορά σε ορισμένες χώρες. Πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν εάν ε, μετρήσουμε το επίπεδο της διαφθοράς σε διάφορες χώρες δηλαδή η πολιτική βούληση, ε, το στερεό και σταθερό νομικό και αστυνομικό πλαίσιο ε, και πολιτικό πλαίσιο και αν υπάρξουν προβλήματα σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά το μείγμα και τον τρόπο με τον οποίο ε, οι εθνικές αρχές αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, ιδίως όσον αφορά αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει ιδίως σε χώρες όπου η πολιτική θέληση δεν ήταν ε, εξίσου ψηλή όπως στο παρελθόν. Τώρα σχετικά με τον ορισμό της διαφάνειας και χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Κίνας αναφέρομαι εις ε, τις ε, ε, αρχικές ε, αρχές και υποθέτω ότι ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την ποικιλομορφία των ε, διαφορών που υπάρχουν σε νομική παράδοση. Πρέπει όμως να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της πολιτιστικής πολυμορφίας και της συμμορφώσεως με τις διεθνείς αρχές οι οποίες περιγράφονται στην σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς και νομίζω ότι με αυτό ολοκλήρωσα. Έτσι έκλεισα και τις συζητήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, κυρία Ματιού θέλει να κάνει μια παρατήρηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ήθελα να απευθυνθώ στην κυρία Βικανάτη. Θέλω να αναφερθώ σε μια υποστολή με την κυρία Γκόμες πήγα στο Αφγανιστάν ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ε μένα με έστειλε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Απλώ για να δούμε αν χρησιμοποιούνται καλά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και μπορώ να σας πω ότι ε, κάπως εξεπλάγει γιατί κάποιοι από τους Αφγανούς συναδέλφους ε, υποπτεύονταν ότι υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς, ε, το ήξεραν ε, δηλαδή ότι υπάρχει διαφθορά στο Αφγανιστάν. Ακούσαμε κάποιους πολιτικούς, αλλά μιλήσαμε και με εκπροσώπους μεγάλων ε, ΜΚΟ και τελικά τι διαπιστώσαμε και αυτό που μας είπαν πάρα πολλές με κυβερνικές οργανώσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και δωρητές είναι ήταν ότι συλλέγονταν ε, από την Παγκόσμια Τράπεζα τα κονδύλια της λοιπόν μάλλον ε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει τόσο διαφθορά γιατί όλα τα ε, συντόνιζε ο με Τράπεζα. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, σας δίνουν λευκή επιταγή ε, τελικά επιτόπου. Δηλαδή, δεν το είπα προηγουμένως, αλλά για αυτό το θέμα ήθελα να σας πω ότι έχετε τεράστια ευθύνη και ηθική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και κάνετε μια πολύ σημαντική δουλειά επ' αυτού, αλλά και επιτόπου και νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνετε και μια δουλειά εκ των υστέρων όταν έχετε εντοπίσει τη διαφθορά. Δηλαδή θα πρέπει να συνομιλείτε και με τα κρατημέλη και με τους δωρητές. Όμως, ε, εντάξει, το ξέρω ότι είναι δύσκολο να ελοπιθεί κάτι τέτοιο, μπορώ να με φανταστώ στη θέση σα, αλλά εγώ νομίζω ότι ε, θα έπρεπε να σκεφτείτε να κλείνετε ίσω και τη βρύση ε, σε τέτοιε χώρε, δηλαδή να μην δίνετε κονδύλια. Δεν είναι εύκολο να το πράξει κανείς, καλό κουράγιο φυσικά, αλλά ε, κάποιοι δωρητές ε, και όσοι δεν εκεί επί τόπου κρύβονται πίσω από τη δική σας εικόνα. Ο κύριο Νιούτον Ντάν θέλει και αυτός να παρέμβει σύντομα. Ε, πολύ σύντομο θα είμαι. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές ε, για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπαν και θα ήθελα να πω ε, πόσο πολύ εντυπωσιάστηκα από την κυρία από το TI ε, που καθόταν εκεί ε, και παράλληλα έγραφε και ανακοινωθέν τύπου για μια άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή και το στη λέγω το είδα στο iPad, μου τρελάθηκα, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ε, κοιτάξτε, έτσι γίνεται σήμερα, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Ρικανατίνη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, θίγεται ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και κατ' ουσίαν μου επιτρέπετε να κάνω μία παρατήρηση που είχα σημειώσει και που ξέχασα να την αναφέρω προηγουμένως. Δηλαδή το ρόλο που έχουμε ε, ως οργανισμός ε, να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Με την έννοια ε, ότι έχουμε τους δικούς μας πόρους και συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις. Εγώ συνεχίζω να τονίζω στους συναδέλφους μου ότι είμαστε ε, δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσιου, ε, διεθνούς οργανισμού, αλλά δημόσιοι υπάλληλοι. Χρησιμοποιούμε κονδύλια φορολογούμενου και φέρουμε ευθύνη για το πώς τα χρησιμοποιούμε. Και δυστυχώς κατά το παρελθόν, τα τελευταία 8 χρόνια, ε, έχουν συμβεί αρκετά πράγματα στην Παγκόσμια Τράπεζα και έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα ολόκληρο τμήμα που ελέγχει πώς ε, χρησιμοποιούμε τους ε, πόρους. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποια υποψία ε, είτε για κάποιο ιδιωτικό φορέα είτε για κάποιο δημοσιογράφο για οποιαδήποτε κονδύλια ε, τα οποία ε, ήταν αντικείμενο κατάχρησης, θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε μία ομάδα εκπαιδευμένων ελεγκτών, ερευνητών ε, που θα παρακολουθήσουν την υπόθεση και μετά υπάρχει μία διαδικασία αξιολόγησης του αποτελέσματος και επιβολής προστήμων και δημοσίευση μαύρου καταλόγου που είναι δημόσιος για όλους και για ιδιώτες και για επιχειρήσεις. Πιέζουμε λοιπόν τόσο πολύ, γιατί αν τελικά είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε αυτό, τότε διαπιστώνουμε ότι και άλλοι, άλλοι φορείς θα συνεργαστούμε και με άλλους φορείς έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει όπως σας είπα ένας ε, μαύρος κατάλογος ε, δημόσιος ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων τραπεζών παραδείγματος χάρη της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε γιατί, γιατί μας καθιστά υπόλογους. Και όπως είπε και ο συνάδελφός μου από την Transparency International, το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει η βούληση, αλλά από όλους. Άρα δηλαδή είμαστε τμήμα εκείνου του ε, κομματιού των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξει η κατάσταση και να δώσουν το καλό παράδειγμα. Γιατί αν ε, δεν, δίνουμε, δεν αλλάξουμε τα, στάνταρτ σε μια χώρα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει διάλογος και να στηρίξει κανείς την αλλαγή σε μια χώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, όσον αφορά τώρα αυτό το μαύρο κατάλογο, υπάρχει μια νέα πολιτική ε, του να είμαστε ανοιχτοί σε οποιασδήποτε μορφή σε έγγραφα και ε, όσον αφορά την πολιτική προσλήψεων ε, στις χώρες, όσον αφορά στις συμβάσεις. Εδώ λοιπόν πραγματικά προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο και λέμε ότι αυτό κάνουμε, παραδείγματο χάρη, ε, στην ακτή ελεφαντεστούν. Ε, αυτό είναι το σχέδιο, αυτά έχουν συμφωνηθεί και όλοι μπορούν να ελέγξουν τους όρους της συμφωνίας, το τι πρέπει να γίνει και πόσα χρήματα δίδονται και μπορούν να επανέλθουν σε μας και να μας βοηθήσουν. Έτσι λοιπόν υπάρχει πολύ βαθύτερη κατανόηση ε, και νομίζω ότι αυτή είναι μια ευρύτερη συζήτηση. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η διαφθορά είναι ένα από τα πράγματα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη και χωρίς ε, την αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν μπορούμε να περάσουμε στην ανάπτυξη. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Ε, αν δεν ε, κινητοποιήσουμε και την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την επιτυχία που επιθυμούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ε, πολλές χώρες μας πλησιάζουν και μας λένε ότι αυτός ο κατάλογος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μήπως μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και εμείς στη δική μας τη χώρα. Έτσι λοιπόν τώρα ε, ξεκινήσαμε αυτό, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις χώρες να συντάξουν ένα τέτοιο κατάλογο ως αποτέλεσμα των ερευνών μιας χώρας έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν ότι παραδείγματος χάρη αυτή η επιχείρηση ή αυτά τα άτομα δεν λειτουργούν μέσα στο ε, ισχύον ε, νομικό πλαίσιο και γι' αυτό έχουν αποκλειστεί για δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. Και πρέπει κανείς να εκπαιδεύσει και τους πολίτες να χρησιμοποιούν σωστά αυτές τις ε, πληροφορίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ πρόκειται για ένα ε, μέσο μακροπρόθεσμο σχέδιο. Ε, Ευχαριστούμε την κυρία Ρακανατίνη, ευχαριστώ τους προσκεκλισμένους μας όχι μόνο που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας, αλλά και επειδή έθεσαν στη διάθεσή μας τις δεξιότητάς τους και την καθημερινή τους δραστηριότητα. Ευχαριστώ την κυρία Μάιερ, τον κύριο Χρυσικό. Εμείς ε, θα ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας τις 3 με κάποιους ε, προσκεκλημένους που θα μας μιλήσουν για την εθνική εμπειρία, για την έρευνα και την πρόληψη της διαφθοράς. Θα τα ξαναπούμε στις 3.